Η διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κέντρα επιχειρήσεων στην Ασία. Θα δώσω το λόγο στο συντάκτη της προφορικής ερώτησης, τον κύριο Μορέιρα δηλαδή, για πέντε λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Την προφορική αυτή ερώτηση την ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και εγώ ω πρόεδρος αυτής τη Επιτροπής θα παρουσιάσω αυτή την προφορική ερώτηση που την έχουν προσυπογράψει και οι κύριοι Κασπάρη, Ρινάλντι, Ζάχερντιλ και Στέρντι. Είναι ε, οι συντάκτες του κειμένου της προφορικής ερώτησης. Το κείμενο της προφορικής ερώτησης είναι γνωστό, δεν πρόκειται να το ξαναδιαβάσω. Θα ήθελα να κάνω κάποια επιπλέον σχόλια. Εδώ μιλούμε για τα ευρωπαϊκά επιχειρηματικά κέντρα στην Ασία που δημιουργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η προώθηση της εμπορίας, ε, του εμπορίου και των επενδύσεων είναι ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και το θέμα αυτό ε, της σύστασης αυτών των επιχειρηματικών κέντρων στην Ασία θα είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν πολύ περιορισμένους πόρους και δεν μπορούν να αφιερώσουν πολλούς στο εμπόριο και στις επενδύσεις. Δημιουργούνται λοιπόν αυτά τα ευρωπαϊκά κέντρα επιχειρήσεων στις τρίτες χώρες για να επιφέρουν μια προστιθέμενη αξία και αυτό γίνεται με υπηρεσίε στήριξη ε, προ ε, τα κράτη-μέλη. εκπρόσωποι των συλλογικών συμφερόντων ε, είναι εκπρόσωποι των συλλογικών συμφερόντων τη Ένωση και προσφέρουν και υπηρεσίε στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Πολλά τέτοια επιχειρηματικά κέντρα ευρωπαϊκά ε, δημιουργήθηκαν στην Ασία. Το 2008 στην Ιδία το πρώτο, 2010 είχαμε στην Κίνα και στην Ταϊλάνδη αντίστοιχη ίδρυση τέτοιων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κέντρων και μάλιστα ε, ε, ανακηρύχθηκε και η ιδέα να δημιουργούνται στο Βιετνάμ, στην Ινδοκίνα και τη Μαλαισία κέντρα στήριξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ευπρόσδεκτη αυτή η πρωτοβουλία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν και ανεπιφύλακτα την υποστήριξε. Αρκεί βέβαια να υιοθετείται μια συνεκτική προσέγγιση και συγκροτημένη. Γι' αυτό ζητήσαμε έναν πιο συγκροτημένο συντονισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και των μελών που φιλοξενούν αυτά τα επιχειρηματικά κέντρα. Μάλιστα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Φεβρουαρίου του 2008, δηλαδή πριν από έξι χρόνια, αναφέρουμε στενότερη συνεργασία με τα εμπορικά επιμελητήρια, με τις ε, εμπορικές οργανώσεις και τις ε, υπηρεσίες προώθηση του εμπορίου που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και, και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των προξενείων ε, και πρεσβειών των κρατών μελών ή άλλες, άλλους φορείς ε, διεθνούς εμπορίου καθώς και τις αρμόδιες ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Αυτά έλεγε το ψήφισμα και επίσης ζητήσαμε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συντονισμού για την παροχή στήριξη προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξασφαλιστεί καλύτερος ο συντονισμός αυτών των δραστηριοτήτων. Προβλέπεται χρηματοδότηση ήδη από το 2012 για τις δράσεις ε, για μια περίοδο που φτάνει μέχρι το 2014. Αναζητούμε λοιπόν μια προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση του εξωτερικού εμπορίου και των επενδύσεων των κρατών μελών. Πέρασαν όμω πολλά χρόνια από την ίδρυση των πρώτων τέτοιων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ε, ε, κέντρων στην Ασία και εν ώψη του μελλοντικού ευρωπαϊκού ανοίγματο και νέων τέτοιων κέντρων και τη μελλοντική ίδρυση, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα απαντήσει κατά πόσο έχει εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των δομών στήριξη. αν ανταποκρίνεται στι προσδοκίε που είχαμε, αν τα αποτελέσματά του είναι ικανοποιητικά και τι μπορεί επίση να γίνει για να βελτιωθεί η δραστηριότητα αυτών των ε, επιχειρηματικών κέντρων και των διαφορών ε, συμπαρομαρτουσών υπηρεσιών στήριξης και πώς, θα εξασφαλιστεί καλύτερο συντονισμός για να ε, εξασφαλιστεί πιο εύρυθμη λειτουργία και των υπαρχών των επιχειρηματικών κέντρων και των μελλοντικών. κυρίως για να εξασφαλιστεί καλύτερη ανάμειξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δεν έχουν ίδιου πόρου και δεν μπορούν ε, να υποφεληθούν ε, από τα κονδύλια των, ε, τα εθνικά. Γι' αυτό και εκεί η παροχή και η στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ανεκτήμητη σημασία. Ευχαριστούμε κύριε Μωρέρο. Ο κύριος Λεβαντόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητά μέλη. Η προφορική ερώτηση αυτή ουσιαστικά αποτελείται από πέντε τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι οι βέλτιστες πρακτικές οι οποίες προσφέρονται μέσω των διμερών ε, επιμελητηρίων και πώς μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα πανευρωπαϊκά κέντρα ιδιαίτερα στην Ασία. Τίθεται λοιπόν ένα θέμα συνοχής με τα υπάρχοντα μέτρα στήριξης αυτών των επιχειρηματικών κέντρων. Η απάντηση είναι ότι τα νέα αυτά κέντρα τα πανευρωπαϊκά της Κίνας και της Ταϊλάνδης μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη ε, λειτουργούν λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες και των κρατών μελών και ενσωματώνοντας όλες τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε αυτές τις χώρες. Αυτό ακριβώς ήταν και η κατευθυντήρια γραμμή για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία την οποία θέλουμε γενικότερα τα πανευρωπαϊκά αυτά κέντρα να αποδίδουν. Το θέμα τώρα της συνδιαχείρισης των υπαρχόντων σωμάτων και υπηρεσιών σε συνέργεια με άλλα μέτρα που υπάρχουν και λειτουργούν ήδη όπως τα help desk, τα επιχειρηματικά δίκτυα στήριξης είναι κάτι ε, που λειτουργεί σαν προϋπόθεση ε, για την σωστή λειτουργία αυτών των πανευρωπαϊκών όπως λέμε κέντρων. Το δεύτερο τμήμα αφορά την κατανομή των πόρων. Υπό το φως του τροπολογημένου κανονισμού, άνω του 50% των διαθεσίμων 76,5 δις για προτεραιότητες 2, στήριξης δηλαδή της επιχειρηματικής συνεργασίας, θα πρέπει να αφιερωθούν σε οκτώ παρεμβάσεις ή επτά άλλωστε μέσω υπαρχόντων επιμελητηρίων. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον καλύπτοντας το 20%. Το θέμα παραγωγής πόρων θα πρέπει να είναι βασικό στόχος της συγχρηματοδότησης αυτών των σωμάτων. Τώρα έχουμε μια νέα γενιά προγραμμάτων για το 2014-2020. Έχουμε το νέο εταιρικό μέσο, το οποίο βασίζεται στα μαθήματα που έχουμε πάρει από το παρελθόν και ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της συνεργασίας με τα άλλα υπάρχοντα μέσα και για τη στήριξη των μικρομεσαίων, ιδιαίτερα που έχουν περιορισμένους πόρους για να διαφημίσουν την παρουσία τους σε αυτές τις απόμακρες για μας χώρες. Το τρίτο τμήμα απαντήθηκε εν μέρη στις δύο προηγούμενες παρατηρήσεις μου. Έχουμε να κάνουμε κάτι το οποίο μας ανησυχεί εδώ. Η προστιθέμενη αξία θα πρέπει να είναι υποστηρίζουν υποστηρίζοντα demand driven, δηλαδή να προκαλείται από τη ζήτηση ε, αυτό είναι κάτι το οποίο περνάει και από την δυνατότητα πρόσβασης στους υπευθύνους αυτών των χωρών, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις. Ενημερωθήκαμε γύρω από τα θέματα αυτά και ένα τμήμα της σύστασης δημιουργεί μια πλατφόρμα συντονισμού για την διεθνοποίηση ε, την καλύτερη δυνατότητα διεθνοποίησης της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ήδη από τις αρχές του 2014 προωθούμε αυτήν την ιδέα. Ε, επανέρχομαι επίσης σε αυτά που είπα στην αρχή της απάντησής μου γύρω από τη συνοχή που θα πρέπει να χαρακτηρίσει τα μέσα αυτά και αυτό είναι προϋπόθεση η οποία ελήφθη υπόψη στο σχεδιασμό των σωμάτων αυτών, των οργανισμών αυτών. Ο υπάρχον κανονισμός τώρα που είναι σε ισχύ τώρα τελειώνει στο τέλος του 2014 για τη δημοσιονομική του στήριξη. Τροπολογήσαμε τον κανονισμό και υπάρχουν νέα μέσα εταιρικά χρηματοδότησης τα οποία βασίζονται στις εμπειρίες του παρελθόντος και αντιμετωπίζοντας ειδικά τις ανάγκες των μικρομεσαίων. Αυτά για την προφορική ερώτηση που αποτελείται από πέντε υποερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τώρα εκ μέρους των πολιτικών ομάδων το λόγο έχει για τρία λεπτά ο κύριος Κάσπαρη. Αξιότιμη Πρόεδρο, αξιότιμη Επίτροπε, η δική μου πολιτική ομάδα, οποτεδήποτε πρόκειται για την βοήθεια και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πάντα στην αιχμή του δόρατος. Και επιθυμούμε να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Θα ήθελα να ε, προβάλλω ιδιαίτερα τις επιτροπές τις οποίες συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες εργάζονται με ιδιαίτερη επιτυχία. Όταν ήρθε η πρόταση να ανοίξει η αγορά για τις μικρομεσαίες χώρες, κυρίως αναδυόμενες χώρες όπως την ε, Κίνα και την Ταϊβάν να υπάρξουν αυτά τα επιχειρηματικά κέντρα. Εμεί την υποστήριξή μα την συναρτήσαμε με το ότι θα πρέπει να τηρούνται κάποιοι όροι. Παραδείγματο χάρη θα πρέπει οι χώρε αυτέ να είναι σημαντικό στόχο για ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, τα κράτη-μέλη να συστήσουν ε, κάποιου οργανισμού, να υπάρχει φιδωλή χρήση των ε, δημόσιων πόρων και επίση θελήσαμε να αποφύγουμε την επικάλυψη εργασιών των ε, υποσύσταση οργανισμών με ήδη υπάρχοντες. Πιστεύω λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι τα τρία κέντρα που ήδη υπήρχαν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένα. Παράδειγμα Ινδία. Η τελευταία έκθεση του επιχειρηματικού κέντρου στην Ινδία που μας βοήθησε και μας εστάλει για την προετοιμασία της σημερινή ε, συζήτησης δείχνει ότι υπάρχουν 17 market issues ε, τα οποία είναι σημαντικά για τα φόρουμ που ασχολούνται με την κατάρτιση πολιτικής. Κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα σε 6 μήνες ε, τέθησαν 17 αιτήματα για πρόσβαση σε αυτό το επιχειρηματικό κέντρο. Δηλαδή 20 εκατομμύρια ευρώ σε 10 χρόνια, άρα 2 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αυτό μας κοστίζει. Στην Ινδία μιλάμε ότι για κάθε αίτημα διατέθηκαν 50.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν είναι αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων και γι' αυτό κύριε Επίτροπε θα ήθελα να απαντήσετε σε αυτό. Η ε, έκθεση του κέντρου στην Κίνα δείχνει βέβαια ότι δέχεται περίπου 100 αιτήματα το μήνα. Το κέντρο στην Ταϊλάνδη κύριε Επίτροπε, το κέντρο αυτό ποτέ δεν πέρασε να ξεπεράσει τα κρατικά προβλήματα. Εν τω μεταξύ στην Μπαγκόγκ ε, γίνονται να κλείσει το κέντρο. Ε, τα κονδύλια μα μας 2 εκατομμύρια ευρώ για το 10 μέχρι 14 απλά εχάθησαν ξαφανίστηκαν. Και όσον αφορά αυτά τα ευρωπαϊκά κέντρα στην Ασία, από ό,τι φαίνεται αγνοήθηκαν βασικές εμπειρίες που είχαν εξαχθεί από ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά κέντρα. Από ό,τι φαίνεται η Κομισιόν που δεν είδε είναι πρόθυμη να διορθώνει λάθος αποφάσεις. Γιατί αλλιώ δεν το καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν κανένα από τα τρία υπάρχοντα κέντρα έστω και για λίγο κατά τη να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις. Ινδονησία, Μαλαισία και εκεί έχουν συσταθεί κέντρα και εκεί υποτίθεται θα συγκεντρώσουμε στοιχεία. Εμεί όμω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, μα ζητήθηκε η γνώμη μα από αυτού και αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπε παρακαλώ να διασφαλίσετε ότι θα δημιουργήσετε πλέον καταστάσει ε, και θα σκεφτούμε όλοι μαζί το πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των κέντρων πριν τα συστήνουμε. Ο κύριο Σεκούτα, παρακαλώ για ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η απόφαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Κέντρων στην Ασία αντασσόταν στην Γενική Ευρωπαϊκή Στρατηγική και την πρωτοβουλία ε, Small Business Act για την υποστηρίξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μόνο 13% των ε, ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων δραστηριοποιείται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να θαρρύνουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που θέλουν να επεκταθούν ε, και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ασία για παράδειγμα, να τι βοηθήσουμε και να αναπτύξουν την ανταγωνιστικότητά του. Η Ασία άλλωστε έχει σημαντικό και ενεργειακό και εργατικό δυναμικό και είναι σημαντικό να έχουμε επιχειρηματικά μας κέντρα και εκεί. Βέβαια, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εκεί πολλές διοικητικές διατυπώσεις ε, και τέτοιες γραφειοκρατικές προκλήσεις. Το θέμα της αποδοτικότητας επίσης που έχει πέσει αρκετά χαμηλά, ιστερεί σε σχέση με τους στόχους μας, ε, είναι μια αρνητική εξέλιξη. Αλλά θα πρέπει να τονώσουμε τον, την ανταγωνιστικότητα και να μην ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ των εμπορικών επιμελητηρίων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα επιτεύγματα των επιχειρηματικών κέντρων και να διορθώσουμε τις αδυναμίες της λειτουργίας τους. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ρευρίσει περαιτέρω το θέμα και να μας ενημερώσει πιο διεξοδικά. Χαίρομαι για την πρόταση των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων του Euro Chambers για μια πράσινη βίβλο με θέμα την οικονομική διπλωματία στην Ευρώπη. Έτσι θα έχουμε μια πιο συγκροτημένη και πανευρωπαϊκή στρατηγική. Ευχαριστώ. Κύριο Ρινάλντι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πιστεύω κύριε Επίτροπε ότι θα πρέπει να βάλουμε λίγη τάξη E Κατανοώ τι δυσκολίε τι οποίε έχουν τα κράτη-μέλη για το συντονισμό των υπαρχουσών δομών. Ε, Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο ελείπει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η συνοχή. Δεν έχει διασφαλιστεί στην παρουσία των επιχειρήσεών μας στην Ασία. Εμείς είδαμε το πώς πηγαίνουν τα πράγματα με επισκέψεις που κάναμε αλλά είδαμε επίσης ότι υπάρχουν και απορίες από αυτά τα οποία είδαμε. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Έχουμε ένα κέντρο στην Ινδία το οποίο κοστίζει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια ευρώ, στην Κίνα 5, στην Ταϊλάνδη 2. Κάθε φορά έχουμε δηλαδή διαφορές πάρα πολύ μεγάλες για το ποιος είναι υπεύθυνο, ποιος συντονίζει, ποια είναι τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν Πολλές φορές, όπως συμβαίνει στην Ταϊλάνδη, συμμετέχει και η Νορβηγία και η Ελβετία, ενώ άλλες φορές όχι. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν μια ολόκληρη σειρά πρωτοβουλειών για την δημιουργία στο Βιετνάμ, στη Μαλαισία, στις Φιλιππίνες, στο Πακιστάν, ίσως σε μια υστερότερη φάση και στο Λάος. Ποιες πρέπει να είναι οι κατευθύνσεις μας λοιπόν για τα επόμενα στάδια. Τα ερωτηματικά είναι ανοιχτά. Πώς θα υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και συμβατότητα στην κατανομή των πόρων. Ε, τις γνωρίζουν τις δομές αυτές οι επιχειρήσεις μας, οι μικρομεσαίες ιδιαίτερα που τις έχουν ανάγκες. Υπάρχουν επικαλύψεις, ποιο είναι το κόστος, η σχέση κόστους-οφέλους. Νομίζω ότι στο τέλος το θέμα γίνεται πάρα πολύ περίπλοκο. Όποιος είναι κοντά σε αυτές τις υπηρεσίες απογοητεύεται περισσότερο από όσο φανταζόταν και υπάρχει πάντως χρόνος για να το διορθώσουμε. Την απουσία του κυρίου Μπουτικόφερ και Σαχράντιλ δίνω το λόγο στον κύριο Πάσκα. Αξιότιμε επίτροπε, Υπάρχουν αυτά τα επιχειρηματικά κέντρα στην Ταϊλάνδη, στην Ινδία και στην Κίνα και τα κέντρα αυτά ε, αντιμετωπίζουν και εξετάζουν διάφορα και διαφορετικού είδους ε, θέματα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι τα κέντρα αυτά χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά κονδύλια και δεύτερον ο ανεξάρτητος ε, έλεγχος έδειξε ότι σε όλα αυτά δυστυχώς υπάρχουν ελλείψεις και λόγω του ότι υπάρχει οικονομική στασιμότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον δεν δικαιούται να διατηρεί αναποτελεσματικές Δομέ δομές. Δομές δηλαδή οι οποίες ε, δεν μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στα, στις επιχειρήσεις. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ελέγξει την ε, αποτελεσματικότητα των κέντρων αυτών στην Ασία και εάν χρειαστεί να προβεί σε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος ε, Στάσνη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ και η δική μου η πολιτική ομάδα ανέκαθεν ήμασταν υποστηρικτές μέτρων πολιτικής που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και πέρα από τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επιχειρηματικά κέντρα στην Ασία είναι ένας τρόπος ε, για να ε, στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν τα κέντρα αυτά πρέπει να λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Δυστυχώς όμως οι τελευταίες αξιολογήσεις κατέδειξαν ότι οι πρωτοβουλίες αυτές ε, δεν ανταποκρίνονται στις δικές μας τις ε, απαιτήσεις. Έχουν τεθεί αρκετά ερωτήματα και πρέπει να σας πω ανησυχούμε για το κατά πόσον οι πρωτοβουλίες που έχουν αληφθεί προσφέρουν ικανοποιητική ε, προστιθέμενη αξία. Ανησυχούμε για το κατά πόσον διαχειρίζονται σωστά οι πόροι, κατά πόσον υπήρξε αρκετή διαφάνεια στην ανάληψη αυτών των πρωτοβουλειών και κατά πόσον τα κέντρα αυτά μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με δικά του έσοδα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η σύσταση νέων επιχειρηματικών κέντρων είναι μια μακροχρόνια διαδικασία και πρέπει να ξεπεραστούν οι αρχικές προκλήσεις. Τα επιχειρηματικά κέντρα στην Κίνα, στην Ινδία και στην Ταϊλάνδη δείχνουν ήδη μια κάποια επιτυχία και νομίζω ότι έχουν και τη δυνατότητα να ενισχύσουν ενισχύσουν τα κοινά μας συμφέροντα. Όμως πρέπει να λογοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κέντρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επίσης να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία και η ενημέρωση αυτά να διατίθενται στις επιχειρήσεις μας έτσι ώστε οι δικές μας επιχειρήσεις όχι μόνο να μπαίνουν στις ασιατικές αγορές αλλά και να ε, ευδοκιμούν σε αυτές. Ευχαριστώ κυρία Κέστιγκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμε επίτρεπε η κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακρογωνιός λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Γιατί οι μικρομεσαίες είναι σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας μεγάλη αξία τους για την διασφάλιση θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω λοιπόν μπορώ να σας πω ότι η δική μου η πολιτική ομάδα στηρίζει ανεπιφύλακτα αυτά τα κέντρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σημειώνουν επιτυχία και λόγω των εξαγωγών τους. Έχουμε μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών χωρίς εμπόδια. Τώρα όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Αν δούμε λιγάκι την αποτελεσματικότητα των κέντρων αυτών θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Έχει λοιπόν φτάσει η στιγμή να διορθώσουμε τα λάθη. Αυτό το ανέφερε ο κύριος Γκασπάρη. Για να είμαστε επιτυχημένοι στις τρίτες χώρες χρειάζεται η τεχνογνωσία, η χρηματοδότηση χρηματοδότηση, βασικές γνώσεις, ε, κατανόηση της ε, τρίτης αγοράς και πρέπει να γνωρίζουμε ε, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, ποια είναι η κατάσταση και πώς είναι δυνατόν να τοποθετηθεί κανείς με τον βέλτιστο τρόπο στην αγορά. Και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα εξωτερικά εμπορικά κέντρα και είναι λυπηρό ότι αυτά δεν λειτουργούν αποτελεσματικά. Ειλικρινά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την πολυτέλεια και νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε τα κέντρα αυτά έχουν μεγάλη αξία για τις ευρωπαϊκές εξαρτήσει. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι κατά πόσον ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις συνέργειες μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ε, μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τη ροή πληροφοριών. Είναι απαραίτητο ε, να υπάρχουν δίκτυα ενημέρωσης και μετά απλά να βρούμε άλλες παράλληλες δομές. Αυτή τη στιγμή ο δρόμος που ακολουθεί δεν είναι σωστός. Βεβαίως καλά αυτά τα επιχειρηματικά κέντρα αλλά πρέπει να πω ότι η επικάλυψη είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε γιατί ε, οδηγεί στο αντίθετο από αυτό που θέλουμε. Η στοχευμένη βοήθεια, αυτό είναι ο στόχος μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τρίτες αγορές. Περνάμε στο Catch the Eye. Μόνο η κυρία Μαγκίνες ζήτησε το λόγο. Κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Στην αρχή τη εβδομάδα. Είχαμε συζήτηση για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Σίγουρα αυτά τα επιχειρηματικά κέντρα θα πρέπει να συζητηθούν και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούσαμε από τον κύριο Κάσπαρη τα προβλήματα. Πολλά θέματα θα πρέπει να διαρευνηθούν. Η ερώτησή μου, κύριε Επίτροπε, είναι εξή. Η ιδέα είναι καλή και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Αλλά τα προβλήματα είναι διαχειριστικά ή διαρθρωτικά γιατί δεν ανταποκρίνονται στο στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκαν αυτά τα επιχειρηματικά κέντρα και πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η δυναμία. Γιατί σίγουρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση από μόνες τους ε, να πάνε στις χώρες αυτές ε, και να δημιουργήσουν εμπορικές διασυνδέσεις. Οπότε αυτά τα εμπορικά ε, επιχειρηματικά κέντρα θα πρέπει να τις βοηθούν και να έχουν προστιθέμενη αξία τι γίνεται με τα κράτη-μέλη και με τα αντίστοιχα ε, δικά του επιχειρηματικά κέντρα. Μήπω υπάρχει μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση, μπορούμε να έχουμε άμυλα και συνεργασία ή συνέργεια. Γιατί έχουμε πολύ χαμηλού ρυθμού οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ε, επιχειρηματικέ ευκαιρίε και εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνε. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν ακούει κανείς τους κυρίους Μορέιρα, Κάσπαρη και τα λοιπά, θεωρεί ότι πράγματι ήταν χρήσιμη η προσπάθεια αυτή ελέγχου την επιδόσεων αυτών των επιχειρηματικών κέντρων. Κανείς δεν αμφισβητεί το σκεπτικό της λειτουργία τους, αλλά είναι σαφές ότι υπογραμμίζονται στις παρουσιάσεις σας αρκετές δυσλειτουργίες και απαιτούνται περαιτέρω έλεγχοι και αναλύσεις κόστους ωφέλους. Συνειδητοποιούμε βέβαια και εγώ πρώτος τους περιορισμούς τους δημοσιονομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης αποτελεσματικής χρήσης των χρημάτων των φορολογουμένων και αυτό κάνω. Ευχαριστώ Επίτροπε. Κλείνει η συζήτηση. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην κοινή συζήτηση για την αλία. Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο μάλλον προφορικές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Γκάλαγκερ. Πέντε λεπτά, ο οποίος όμως δεν είναι εδώ. Οπότε